Bene, ciao. Non so come si fa qua. Bene, prego. Ας ξεκινήσουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε. Φορέστε τα ακουστικά σας. Και όσοι είναι όθοι, ας καθίσουν παρακαλώ, για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας δύο σημαντικούς εκπροσώπους της Ιταλικής κυβέρνησης, της Προεδρίας δηλαδή, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εξάμεινο αυτό. Παρακαλώ, μην μιλάτε εκεί στο βάθος γιατί δημιουργείται βασάρια. Έχουμε μαζί μας τον Υπουργό κ. Ντάριο Φραντσασκίνη και τον Υφυπουργό κ. Τζακομέλη που θα παρουσιάσουν τις προτεραιότητες της Ιταλικής Προεδρίας. Θα προχωρήσω γρήγορα στην έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Υπήρξαν κάποιες αλλαγές όπως βλέπετε στο προβλεπόμενο στο σημείο 4 στις ακροάσεις. Όπως βλέπετε δεν είναι παρούσα σήμερα, δεν θα είναι παρούσα σήμερα, αλλά αύριο στις 11 υπουργό στις 10 διορθώνει πρόεδρος, η υπουργός κυρία Τζανίνη, Στεφάνια Τζανίνη, Υπουργό ε, Παιδείας, γιατί σήμερα στη Ρώμη υπήρχε η Σύμβουλο Υπουργών για τη μεταρρύθμιση των σχολείων. Θα έρθει αύριο. Αργότερα θα έρθει ο Υφυπουργό κύριος Μπόμπα υπεύθυνο για τις πολιτικές για την νεολαία που θα μιλήσει για το θέμα του αθλητισμού. Αν συμφωνείτε, καταγράφουμε την αλλαγή και προχωρούμε. Παρακαλώ να εγκρίνουμε τα πρακτικά τη συνεδρίας τη 7 η Ιουλίου. Αν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις, θεωρήσω ότι έγινε. Έγιναν δεκτά. Προχωρούμε στο επόμενο σημείο. Εγκρίνονται τα πρακτικά της 7 η Ιουλίου, όπως σας είπα. Τελευταία ανακοίνωση. Να σας ενημερώσω ότι η συνεδρίαση ακούγεται σε live streaming άρα μπορεί να το, την ακούσουν οι πάντες. Και έχουμε διερμηνία σε πολλές γλώσσες, μεταξύ των οποίων και τα ελληνικά. Θα περάσουμε στο σημείο 4, παρουσίαση της Ιταλικής Παιδείας του Συμβουλίου. Είναι σημαντική ευκαιρία αυτή που έχουμε ως Επιτροπή Πολιτισμού που όπως γνωρίζετε ασχολείται με πολλά θέματα, αθλητισμό, νεολαία, η πολιτιστική διάσταση στη συνεργασία με τρίτες χώρες, μέσα ενημέρωσης, οπτικοακουστικά μέσα. Να ευχηθώ λοιπόν κάθε επιτυχία στην Ιταλική Προεδρία που είχε κάπως ε, πιεσμένο χρόνο γιατί ήταν σε μια περίοδο που ούτε η Επιτροπή είχε ξεκινήσει, εμείς είχαμε μόλις ξεκινήσει τη θητεία μας, ήταν και το καλοκαίρι στη μέση. Θεωρώ ωστόσο ότι είναι μια στρατηγική σημασία προεδρία, καθώς ξεκινάμε το νέο κοινοβούλιο, με την νέα περίοδο, εύχομαι, των ευρωπαϊκών πολιτικών και αύριο την έγκριση των πολιετών προγραμμάτων, τα οποία είναι πλάκη πολύ και η Επιτροπή μας ο προγραμματισμός για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την δημιουργική Ευρώπη, το Εράσμος, οι πολιτικές για τους νέους, η Ευρώπη των πολιτών και μια σειρά άλλων πολιτών προγραμμάτων. Θα δώσω λοιπόν αμέσω το λόγο στον κύριο Φραντσεσκίνη για να μας παρουσιάσει τις προτεραιότητες της Ιταλικής Προεδρίας. Ο κύριος Φραντσεσκίνη είναι υπουργό Πολιτισμού, Τουρισμού και Πολιτισμικών Αγαθών είχε πάει και στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, γι' αυτό καθυστέρησε λίγο. Τον συγχωρούμε, γιατί ξέρετε δεν μπορεί να είναι πανταχού παρόν. Θέλω να ζητήσω ωστόσο από τον κύριο Φραντσισκίνη να μας πει εξ αρχής ένα πράγμα. Γνωρίζουμε ότι η Ιταλική κυβέρνηση και η Ιταλική Προεδρία θέλουν, το έδειξαν ήδη, θα μας το πείτε, να ε, δοθεί μεγαλύτερη έμφαση από ό,τι στο παρελθόν στην πολιτιστική πολιτική την πολιτιστική κληρονομιά, ηλική και άειλα, την ψηφιακή πρόκληση ε, και τα θέματα της ολοκληρωμένης προσέγγισης του πολιτισμού με άλλες δράσεις όπως τον τουρισμό, Φερρυπίν, ή οικονομικά ζητήματα όπως τα, δικαιώματα, τα συγγραφικά δικαιώματα. Περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν τους, ώστε η οικονομικα ζητηματα οπως τα δικαιωματα τα συγγραφικα δικαιωματα περισσοτερο απο οτι στο παρελθον του ωστε η στρατηγικη για την Ευρώπη 2020 να αλλάξει, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στα θέματα αυτά σε μια νέα φάση ανάπτυξης και ε, πρόοδου. Θα ήθελα να ρωτήσω να υπάρξει σαφής δέσμευση και της Ιταλικής Προεδρίας στο θέμα, το λεπτό θέμα που θα εξετάσουμε αύριο, την έγκριση του προπολογισμού το 2015 της Επιτροπής. Εγώ είμαι η συνεισηγήτρια για τον πρώτο προπολογισμό του επομένου έτους και πρέπει να σας πω ότι ανησυχούμε ιδιαίτερα λόγω των περικοπών που ξέρω ότι προσπάθησε να περιορίσει η Προεδρία αλλά παραμένει διότι πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει συμμαχία με το Κοινοβούλιο γιατί είμαστε συν νομοθέτες ώστε να αποκατασταθούν ε, τα κονδύλια για τον πολιτισμό ιδίω να μπορέσουν να ελοπιθούν τα προγράμματα που εγκρίνουμε. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε. Σας δίνω το λόγο κύριε Υπουργέ για τα θέματα τώρα που έχουν να κάνουν με το οπτικοακουστικά μέσα και τα ICT. Έχει δώσει το λόγο μετά στον κύριο Τζακομέλη που είναι υφυπουργό ανάπτυξης με αρμοδιότητες της τηλεπικοινωνίας και της συχνότητε. που είναι, τονίζω, στο κέντρο των μελλοντικών πολιτικών. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Καταρχάς, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Αλλά στην προηγούμενη επιτροπή που είχα πάει για τον τουρισμό είχα πολλές ερωτήσεις και χρειάστηκε να ξεπεράσουμε τον χρόνο που, είχα, που είχε προβλεφθεί για να μην αφήσω αναπάντητα τα ερωτήματα που είχαν τεθεί. Πιστεύω ότι το εξάμεινο της Ιταλικής Προεδρίας έχει το όριο του εξαμήνου αλλά και την ευκαιρία να τον περιορισμό αλλά και την ευκαιρία να δουλέψει με ένα νέο κοινοβούλιο και με μια κομισιόν που ξεκινά μόλις τη θητεία της. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να κάνουμε μαζί μια νέα αρχή στο θέμα του πολιτισμού μαζί με το Κοινοβούλιο ε, να μπορέσουμε να διοθετήσουμε κάποιες βασικές αξίες που σχετίζονται με μια μεγάλη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Όλοι εμείς που είμαστε εδώ παρόντες αποφασίζουμε κατά κάποιο τρόπο για τον τομέα του πολιτισμού. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι χρειάζεται να σας ε, να πιστούμε αμοιβαία για το κεντρικό χαρακτήρα που πιθανώς έχουν οι πολιτιστικές πολιτικές για την ανάπτυξη της Ευρώπης χρειάζεται να πείσουμε τους άλλους που λαμβάνουν αποφάσεις εκτός πολιτισμού για το ότι ο τομέας αυτός είναι κεντρικής, κομβικής σημασίας για να αποκτήσει ως Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικές κυβερνήσεις την επίγνωση ότι η πολιτιστική μας κληρονομιά, η ομορφιά της κληρονομιάς μας, η σπουδαιότητα της πολιτιστικής, της ιστορίας, η σπουδαιότητα της δημιουργικότητας και το, της πολιτιστικής βιομηχανίας που σχετίζεται με τη δημιουργικότητα από κοινού αποτελούν το μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ευρώπης στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Το χαρτί στο οποίο θα πρέπει να, θα πρέπει να επενδύσουμε στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα που θα καταστήσει την Ευρώπη ισχυρή και θα επιτρέψει να γίνει παράγοντας ανάπτυξης. Η επένδυση λοιπόν στην προστασία της κληρονομιάς, στην, ε, η επένδυση στο ταλέντο των δημιουργών μας, όλων των επαγγελμάτων που σχετίζονται με τη δημιουργικότητα μπορεί να αποτελέσει πραγματικά το ατού με το οποίο θα κερδίσουμε σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο σε όπου σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις περιοχές του κόσμου θα πρέπει να εντοπίζουμε κάθε φορά τι, σε τι είμαστε καλύτεροι, σε τι είμαστε πιο ανταγωνιστικοί και σε αυτό να επενδύουμε. Είναι προφανές ότι ήμουν στον τουρισμό προηγουμένω και όπω καταλαβαίνετε και ο πολιτισμό και ο τουρισμό συνδέονται στενά. Οι επενδύσεις στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, στη δημιουργικότητά μας, είναι προϋπόθεση για να τραβήξουμε νέο τουρισμό, άρα να έχουμε οικονομική ανάπτυξη. Είναι όμως και προϋπόθεση για να προσελκύσουμε επενδύσεις, γιατί οι επενδύσεις γίνονται ανά τον κόσμο, λαμβάνοντας υπόψη πολλές παραμέτρους. Σε κάποιες περιπτώσεις το κόστος της εργασίας, σε κάποιες περιπτώσεις το που βρίσκεται η επένδυση, σε άλλες η εξαιρετική ικανότητα που παρέχει η Ευρώπη να προσφέρει ποιότητα, ομορφιά, όρους δηλαδή προσέλκυσης επενδύσεων από την υψηλότερη βαθμίδα των επενδυτών. Σε αυτό προστίθεται το ότι ο πολιτισμός είναι προφανώς το ισχυρότερο εργαλείο για να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή ταυτότητα, την κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα και για να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ της ε, προάσπισης της εθνικής ταυτότητας και των, διαφορετικών εθνικών ταυτοτήτων με την οικοδόμηση μιας κοινή ευρωπαϊκής ταυτότητας. Ο πολιτισμός είναι το εργαλείο για να αντιμετωπίσουμε την, το, το, το διώνυμο αυτό, αλλά και για να καταστήσουμε τον κόσμο πιο ωραίο πιο έξυπνο όταν χρειάζεται να ε, αντιπαρατεθούμε με, νέες, με νέους πολιτισμούς, με νέες κουλτούρες της μετανάστευσης που ο αιώνας αυτός θα μας φέρει μπροστά. Η αναθεώρηση λοιπόν της στρατηγικής Ευρώπη 2020 μας προσφέρει την ευκαιρία να ξεκινήσουμε αυτή την ενάρετη πορεία αναδεικνύοντας τον, ε, τις δημιουργικές επιχειρήσεις του πολιτισμού και τον πολιτισμό και η Προεδρία θέλει να προωθήσει ε, αυτό το θέμα στη συζήτηση στο Συμβούλιο. Θα δεσμευτούμε λοιπόν για να αντιμετωπίσουμε και να αξιοποιήσουμε εξ αρχής ε, την έννοια της, του εγκάσιου χαρακτήρα των πολιτιστικών πολιτικών. Διπολιτιστικές πολιτικές μπαίνουν σε πολλούς τομείς. Ε, συνοχή, περιφερειακή ανάπτυξη, τουρισμό, φορολογία, εκπαίδευση, έρευνα. Πρέπει να κάνουμε τον πολιτισμό, την πολιτιστική μας κληρονομιά, ένα όπλο που θα κερδίζει και να το αναδείξουμε. το πολιτιστικό ζήτημα που ήταν αντικείμενο και των συναντήσεων των Υπουργών Πολιτισμού στην τελευταία συνάντηση επί ελληνικής προεδρίας με, διάφορο, με διάφορη σύνδεση αλλά με κοινό τρόπο δόθηκε στην Επιτροπή στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων με τη ΣΥΠΑ η εντολή να διατηρηθεί η εξαίρεση του πολιτισμού. Πρέπει να εξηγήσουμε σε εμά πρώτα ότι το μέτρο αυτό δεν είναι προστατευτικό μέτρο. Εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε, δεν θέλουμε να προστατεύσουμε με την πολιτισμική εξαίρεση, εξαίρεση τους, πολιτικούς και την παραγωγή μας. Θέλουμε να πείσουμε τους διαπραγματευτές της είπα αύριο όλο τον κόσμο ότι η πολιτιστική εξαίρεση σημαίνει να μην δίνουμε τον, να μην μετατρέψουμε τον πολιτισμό και ό,τι συνδέεται με τον πολιτισμό σε ε, ένα εργαλείο που υπακούει μόνο στην λογική της αγοράς. Δεν μπορεί να αγνοηθεί αλλά δεν μπορεί η οικονομία να είναι ο μόνος, η μόνη παράμετρος του πολιτισμού. Αυτό είναι η βαθύτερη σημασία της πολιτιστικής εξαίρεσης. Κατά συνέπεια, ε, ο πολιτισμός στο κέντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής, μοντέλο διακυβέρνησης που μοιράζονται το δημόσιο και οι ιδιώτες. Προσπαθούμε να ετοιμάσουμε ένα νέο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Μερίσης Διάταξης του Πολιτισμού μετά το 2014 από το 2015 και μετά δηλαδή, όταν θα, που θα εγκριθεί στην Σύνοδο Κορυφής των Υπουργών το Νοέμβριο του 2014 και θέλουμε το πρόγραμμα αυτό να είναι ένα πρόγραμμα για τον πολιτισμό κοινά αποδεκτό. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το ευαίσθητο ζήτημα της ψηφιακής επανάστασης. Τα θέματα που συνδέονται διαφορετικά θέματα που συνδέονται όμως με την πνευματική ιδιοκτησία, την αντιμετώπιση της πειρατείας και την φορολογική ισορροπία. Είναι προφανές στο πλαίσιο αυτό ότι τα θέματα αυτά είναι θέματα που όλο και λιγότερο θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν σε εθνικό επίπεδο από εθνικές πολιτικές. Ενώπιον παγκοσμίων φαινομένων που δεν καταλαβαίνουν τις αποστάσεις, δεν καταλαβαίνουν τα σύνορα, χρειάζεται να υπάρχει ένα επίπεδο αντιμετώπισης πιο πάνω από το εθνικό. Ιδίω το θέμα που αφορά τον κλάδο μας. Είναι ένα ευαίσθητο θέμα που πρέπει να δούμε διεξοδικά και με ανοιχτό τρόπο. Και προφανώς η συζήτηση με το Κοινοβούλιο θα έχει σημαντικό ρόλο τη σχέση μεταξύ copyright και της ψηφιακής εποχής. Η αντιπαράθεση μεταξύ της σωστής, του σωστού αιτήματο ελευθερίας στην πρόσβαση στο περιεχόμενο που προκύπτει από το ίντερνετ όταν συναντιέται με το δικαίωμα των συγγραφέων να αναγνωρίζεται θεμητά το δικαίωμα αμοιβή για τη δουλειά τους. Διότι ο δημιουργός είναι αυτός που εξασφαλίζει την το δικαίωμα του δημιουργού εξασφαλίζει την ελευθερία της δημιουργίας. Το θέμα αυτό ουδέποτε μέχρι σήμερα είχε βρεθεί σε τόσο... τα, δύο ζητήματα δεν είχαν ποτέ βρεθεί σε τόσο ε, έντονη σύγκρουση μεταξύ τους. Πρέπει να προσπαθήσουμε να ε, διαμεσολαβήσουμε με δίκαιο τρόπο. Η Προεδρία κατόπιν θα ασχοληθεί με θέματα που βρίσκονται η υποεξέλιξη η πρωτοβουλία Ευρωπαϊκά που είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα που ασχολείται με την πολιτική κληρονομιά και επιτρέπει σε και μεγαλύτερο αριθμό πολιτών να έχουν πρόσβαση στην ευρωπαϊκή πολιτική κληρονομιά, να αναπτύξουν νέε μοντέλα δημιουργική οικονομία και επιχειρηματικότητα. Μεγαλύτερη ενσωμάτωση λοιπόν μεταξύ ερευνητικών υποδομών και ψηφιακών υποδομών κάτι που πρέπει να υπογραμμίσω και που τονίζει η UNESCO ότι ονομάζονται ε, της ανθρωπότητας που είναι η προστασία ενός κράτου ή μιας, κράτους ή μιας δομής που δεν μπορεί να αγνοηθεί από την υπόλοιπη ε, ανθρωπότητα. Η... Πιστεύω ότι τούτο και τέθηκε στην τελευταία συνάντηση του Συμβουλίου Υπουργών Πολιτισμού είναι πραγματικότητα, θα πρέπει να μπορέσουμε να φανταστούμε μορφές παρέμβασης σε περίπτωση φυσικών καταστροφών που πλήττουν την κληρονομιά και που παρέχονται όχι με εθνικές μορφές αντιμετώπισης αλλά με ευρωπαϊκές μορφές αντιμετώπισης, κυρίως οικονομικής. Ένα άλλο μοντέλο είναι να επενδύσουμε στην κινητικότητα των ε, καλλιτεχνών ένας άλλος τρόπο δημιουργία δηλαδή ευρωπαϊκής ηθαγένεια και αξιοποίησης του ταλέντου των νέων της Ευρώπη μέσω ενός συστήματος σπιτιών καλλιτεχνών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με τον εντοπισμό, μια ιδέα που θέλουμε να δουλέψουμε, ενός προγράμματος που δεν θα είναι ένα Εράσμους αλλά θα μοιάζει με τη, στη φιλοσοφία του με το Εράσμους που θα βοηθά στο μέτρο του δυνατού την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ νέων που δουλεύουν στον τομέα της, στον τομέα πολιτικής κοινωνίας σε διάφορες χώρες ε, της Ένωσης, ενώ ταυτόχρονα θα υπάρχουν ανταλλαγές μεταξύ μουσείων, ε, αρχαιολογικών ε, και αρχαιολογικών χώρων, κάτι που θα πρέπει την δυνατότητα ανταλλαγών, γιατί το πιο σημαντικό που πρέπει και μπορούμε να κάνουμε είναι να επενδύσουμε στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Να επενδύσουμε στους νέους, σε κάθε επίπεδο. Θα αύριο θα έχει την ακρόαση και με την Υπουργό Παιδείας και Πανεπιστημίων. Να επενδύσουμε για να μπορέσουν οι νέοι να καταλάβουν καλύτερα την ανάγκη πολιτισμού σε κάθε επίπεδο. Ό,τι μπορεί να είναι χρήσιμο και ένα άλλο μεγάλο θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε στην ψηφιακή εποχή είναι η προσαρμογή του ΦΠΑ μεταξύ του ηλεκτρονικού βιβλίου και του βιβλίου σε χαρτί. Κάτι που πρέπει να αποφασιστεί επίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και οι πολιτικές ε, αδελφοποίησης που επιτρέπουν την, το να μοιράζονται εμπειρίες. Στην Επιτροπή Τουρισμού ε, δημιουργήθηκε η, η ανάδειξη των ευρωπαϊκών δρόμων που μέσω πολλών ευρωπαϊκών χωρών αποτελούν εργαλείο όχι μόνο προσέλκυσης τουριστών σε περιοχές που είναι τουριστικές, δηλαδή πρωτεύουσε ε, ή τουριστικά κέντρα, αλλά που βοηθούν να προχωρήσει ο τουρισμός και αλλού με την παροχή βοήθειας από χώρες που έχουν τουριστική εμπειρία σε χώρες με μικρότερη τουριστική εμπειρία. Αυτοί οι δρόμοι, αυτές οι διαδρομές που μπορεί να είναι διαδρομές με τα πόδια, με τρένο, με ποδήλατο έχουν μεγάλη αξία σύνδεσης στις 9 Σεπτέμβρη, στα πλαίσια του εξαμήνου του... της Προεδρίας, θα υπάρξει στις Βρυξέλλες μία έκθεση ε, για την πόλη της Σιένα. Η δύναμη της Σιένα στην αναγέννηση ήταν ότι βρισκόταν στην Βία Φραγκίτζενα, δηλαδή τον δρόμο που από τη, από τη Βόρεια Ευρώπη οδηγούσε προς τους Αγίους Τόπους μέσω των μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων. Ήταν το σημείο ε, ήταν σημείο, ήταν σταυροδρόμι, σημείο συνάντησης και διαλόγου μεταξύ των διαφόρων πολιτισμών, των διαφόρων κουλτουρών, ούτως ώστε η ανάδειξη αυτών των διαδρομών μπορεί να αποτελέσει ένα μεγάλο εργαλείο γνώσης και εν, ενοποίησης, όπως πρέπει να βοηθήσουμε και άλλους τομείς που σήμερα αντιμετωπίζουν κίνδυνο περιθωριοποίησης, Φερρυπίν, η πρόταση των μικρών ε, κινηματογραφικών αιθουσών, των ε, την, λογοτεχνική, με, την αξία της λογοτεχνικής μετάφρασης. Να φανταστούμε μια ε, ε, ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτά τα πράγματα και είναι κάτι πάνω στο οποίο δουλεύουμε και ελπίζουμε μετά την Ιταλική Προεδρία να ολοκληρωθεί αλλά θέλουμε να υπάρξει ε, μια διάσκεψη της, ε, όλων των φορέων της, της ευρωπαϊκής πολιτιστικής βιομηχανίας, όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι στον πολιτισμό που έχουν καταλάβει τον κεντρικό, τον κομβικό ρόλο που μπορεί να έχει μια επένδυση στον τομέα αυτό, θα πείσουν άλλους υπεύθυνου ε, για τον κεντρικό χαρακτήρα του κλάδου. Και εδώ ιδίω σε σχέση με την ενσωμάτωση, με το συσχετισμό κουλτούρας, πολιτισμού και τουρισμού. Και δεν το λέω αυτό επειδή ε, το χαρτοφυλάκιό μου έχει αυτά τα δύο, αλλά γιατί είναι προφανές ότι ο τουρισμός από την Ευρώπη, ο τουρισμός στην Ευρώπη, συγγνώμη, ε, έρχεται κυρίως λόγω της μεγάλης πολιτιστικής προσφοράς της Ευρώπης. Το ταξί, ο λόγος του ταξιδιού είναι κυρίως αυτός. Και σήμερα η επιλογή του ταξιδιού είναι η επιλογή του να πάω στην Ευρώπη, όχι να πάω σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Ίσως αυτή η ευκαιρία να προκύψει μια φορά στη ζωή κάποιου. Άρα αυτό ο κάποιο δεν θα πάει σε μια χώρα αλλά στην Ευρώπη. Εμεί λοιπόν αυτός, θεωρούμε ότι αυτό είναι ακόμα λόγο για να δουλέψουμε και να παλέψουμε για την ε, ενσωμάτωση του τουρισμού και του πολιτισμού. Για το λόγο αυτό κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα οργανώσουμε στην Άπολη μια γενική συνάντηση για τον, ένα ευρωπαϊκό φόρουμ για τον τουρισμό 29-30 Οκτωβρίου, όπου θα καλέσουμε όχι μόνο υπουργού τουρισμού, αλλά και υπουργού πολιτισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση και όλου του εμπλεκόμενου στον κλάδο, ούτω ώστε να δούμε πώ θα μπορέσουμε να ενοποιήσουμε ή να φέρουμε πιο κοντά του δύο αυτού προπολογισμού, του δύο αυτού, ε, τι δύο αυτέ κατηγορίε. Για τον προπολογισμό τώρα που μου ζήτησε η πρόεδρο, το κοινοβούλιο μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο όχι για το νούμερο, αλλά για το μήνυμα που θα περάσει για τον πολιτισμό. Και ως παιδεία θα προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε στην εξέβρεση μιας λύσης στον τομέα αυτό. Αμέσως δίνω το λόγο στον κύριο Τζακομέλη. Ξέρω ότι η Επιτροπή μας ενδιαφέρεται και για όλα τα θέματα της ψηφιακής ε, πρόκλησης που είναι ένα σημαντικό θέμα το λόγο έχει ο κ. Τσακουμέλη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Προφανώς ο οπτικοακουστικός κόσμος ε, εμπλέκεται σε μια βαθιά αλλαγή και πρέπει να αντιμετωπίσει η δυσκολία που αντιμετωπίζει είναι ότι αλλάζει η σύγκληση, αλλάζει ο τρόπος διανομής, κατανάλωσης του τηλεοπτικού και κινηματογραφικού περιεχομένου η ψηφιακή επανάσταση επιβάλλει να λάβουμε υπόψη τελείως διαφορετικές πραγματικότητες σε σχέση με αυτές που είχαμε συνηθίσει. Ενώπιον αυτών των εξελίξεων η Ιταλική Προεδρία θεωρεί ότι βεβαίω είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις του ώστε η Ευρώπη να είναι μια ενιαία ψηφιακή αγορά, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορεί η Ευρώπη να είναι μόνο αγορά, αλλά και ένα πολιτικό και θεσμικό υποκείμενο ικανό να παρέμβει και να αλλάξει τις προϋποθέσεις για να αποφύγουμε τον κίνδυνο που προφανώς η νέα σύγκληση επιβάλλει. Άρα πρέπει να υπάρχουν προσπάθειες να αντιμετωπίσουμε την σύγκληση μόνο σε εμπορικό ε, σε, από εμπορική οπτική γωνία και να θεωρήσουμε ότι το διαδίκτυο δεν μπορεί να είναι μόνο ένας χώρος εμπορικής δράσης. Ε, πλέον αντιμετωπίζεται ως μια προβολή του εαυτού σου, ένας χώρος ελευθερίας, ένας χώρος έκφρασης, συνάντησης και άρα υπάρχει ανάγκη να προστατεύεται υπό τον όρο αυτό της ελευθερίας και της ευκαιρίας που παρέχει. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για την σχέση με την παραγωγή που είναι προϊόν του πολιτισμού, την κινηματογραφική παραγωγή, την οπτικοακουστική παραγωγή και τις συναφείς δραστηριότητες. Εμείς συμφωνούμε βεβαίως με την επιλογή της πολιτιστικής εξαίρεσης που ανέφερε ο Υπουργό κ. Φραντσεσκίνη. Είμαστε βαθιά πεπισμένοι για την αναγκαιότητα αυτής της επιλογής. Βεβαίως όλοι έχουμε επίγνωση ότι η επιλογή αυτή δεν μπορεί να λειτουργήσει μακροπρόθεσμα, αλλά μόνο να κερδίσουμε χρόνο, κάτι που επιβάλλει κατά την άποψή μα στι ευρωπαϊκέ κυβερνήσει, την εξή πρόκληση ή και την εξή δυνατότητα, την ικανότητα αναδιοργάνωση του πολιτισμού ω προ τον πολιτικό ρόλο, τον κανονιστικό ρόλο, τον ρόλο των θεσμικών οργάνων, αλλά και την οργάνωση ολόκληρη ενός κλάδου κάτω από τις νέες παγκόσμιες συνθήκες τα στοιχεία της πολιτιστικής παραγωγής στο διαδίκτυο ε, έχουν αμερικανική προφορά, αλλά παρέχουν και το αποτέλεσμα του, αποτέλεσμα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Γι' αυτό σε ένα ε, σε ένα, ε, ε, ένα συμβούλιο που έγινε στο Μιλάνο, άτυπο συμβούλιο στο Μιλάνο για την διακυβέρνηση του ίντερνετ, αποφασίσαμε ότι η Ευρώπη πρέπει να μπορεί να μιλήσει ε, με μία φωνή στην ψηφιακή, στον ψηφιακό κόσμο για να θέσουμε ενώπιον τον είπα την ευρωπαϊκή θέση. Ξέρουμε πολύ καλά πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος γιγάντων του διαδικτύου, αυτό που λέμε over the top πρόκειται για, οργανο, οργανισμούς που, που σηματοδοτούν εμπορικά, πολιτιστικά, οικονομικά το πεδίο της πολιτιστικής και οικονομικής πραγματικότητας. Αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Κρατώντας βέβαια την αρχή που και η Επιτροπή ε, υπογραμμίσει την ουδετερότητα του διαδικτύου, το net neutrality και με σεβασμό της ισότητας ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων χρηστών της πλατφόρμας του διαδικτύου και εκμεταλλευόμενοι την ικανότητα που έχουμε να μπορούν όλοι οι εμπλεκόμενοι να, αντιμετω... με τον ισότιμο τρόπο. Πρόκειται βεβαίως για παραγωγές που είναι καρποί εθνικών πραγματικοτήτων. Εμείς λοιπόν πρέπει να ζητήσουμε να υπάρχει μία σχέση με τους θεσμούς και τον πολιτισμό της κάθε χώρας στους, από τους ε, μεγάλους χειριστές πλατφόρμας που θα επιτρέπουν ίση αντιμετώπιση του κάθε, κάθε εμπλεκόμενου, οικονομικά εμπλεκόμενου στο διαδίκτυο η απόφαση του Federal Communication Commissioner, τον ΗΠΑ, προσανατολίζεται προς την δημιουργία μιας συμφωνίας μεταξύ χρηστών και, και οργανώσεων, ε, οργανισμών τηλεπικοινωνιών. Αυτό είναι ένα γεγονός που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Προφανώς κάθε συμφωνία είναι θετική, αλλά εμείς πρέπει να προσέχουμε ούτως ώστε η συμφωνία μεταξύ μεγάλων ομίλων δεν θα παίξουν το ρόλο που, θα, που κανονικά θα έπρεπε να παίξουν τα θεσμικά όργανα των κρατών. Εμείς δεν μπορούμε να αφήσουμε ε, το διαδίκτυο να λειτουργήσει βάση των αποφάσεων, ε, των οικονομικών αποφάσεων των μεγάλων ε, επιχειρήσεων του διαδικτύου. Και εδώ υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία για την Ευρώπη με τις διάφορες οδηγίες, π.χ. η οδηγία για την ψηφιακή ενιαία αγορά και άλλες, για να παρέμβουν και να παίξουν ρόλο και κάτι που θεωρώ σημαντικό είναι ότι πιστεύω ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε και νομίζω το είδατε στην επιτροπή σας πρόσφατα την οδηγία Μέντια. γιατί από την άποψη αυτή συμφωνώ με τις θέσεις αν τις θυμάμαι σωστά το ψήφισμα Κόμεμπερ του Ιουλίου του 2013 που κατά βάση έθετε ακριβώς το θέμα του ότι μπροστά στην σύγκληση που, που εξελισσόταν το νομοθετικό πλαίσιο ήταν ανεπαρκές και απαιτούσε μια πιο διεξοδική και όχι μόνο ε, οικονομική ανάλυση της κατάστασης. Πιστεύω ότι μπροστά μας έχουμε μια μεγάλη πρόκληση. Την ψηφιακή επανάσταση που ζητά και νομοθετική παρέμβαση, αλλά κυρίως πολιτιστική. Εμείς έχουμε μπροστά μας αυτή την επιλογή. Και εδώ θέλω να κλείσω. Μπορούμε να επιτρέψουμε το έργο το δικό μας, τόσο εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο, ε, μπορούν, μπορεί να είναι ε, έργο παρέτησης υπέρ των εμπλεκομένων στο διαδίκτυο ή από την άλλη να δείξουμε ότι η σύγκληση ε, δίνει ευκαιρίες για όλου να το αποφασίσουμε αυτό και να μην δημιουργήσουμε οικονομικά εμπόδια που θα στηρίζονται στα συμφέροντα των μεγάλων οικονομικών πραγματικότητων, αλλά όλων. Αυτή είναι και, αυτός είναι και ο στόχος μας. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ για τις δύο παρεμβάσεις σας. Θέλω να ακούσω τις ε, παρεμβάσεις. Ε, Καμερέμπερ, Διβάτσκα και Αντινόλφη. Κάποιοι άλλοι θέλουν το λόγο. Η κυρία Καμερέμπερ πρώτα. Ευχαριστώ θερμά κύριε, κύριε Υπουργή. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα επειδή με σαφήνεια είπατε πόσο ο πολιτισμός έχει σημασία, μεγάλη σημασία ε, για την Ιταλική Προεδρία και βέβαια και το Κοινοβούλιο είχε ε, τονίσει ότι θα πρέπει να εξαιρεθούν ε, όλα τα οπτικοακουστικά μέσα από το TTIP ότι, και το είχαμε τονίσει αυτό. Ένα λεπτό για να φτιάξει ο κύριος υπουργό τα ακουστικά του που δεν λειτουργούν. Είναι εντάξει, λειτουργούν, εντάξει, ακούτε, ωραία, ωραία. Λυπάμαι, θα ξαναρχίσω. Κύριοι Υπουργοί, Ευχαριστώ θερμά για τις εισηγήσεις σας και ευχαριστώ ιδιαίτερα επειδή τονίσατε με μεγάλη σαφήνεια πόσο σημαντική είναι η, πολιτιστική, ε, η εξαίρεση των πολιτιστικών θεμάτων από την συμφωνία TTIP. Ξέρω η Ιταλική κυβέρνηση και στο Συμβούλιο έχει τον ΙΣΙ έχει πιέσει ιδιαίτερα να εξαιρεθεί αυτός ο τομέας από το διαπραγματευτικό πακέτο αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τονίσει ότι πρέπει να εξαιρεθεί όχι μόνο από τα πολιτιστικά θέματα αλλά και από τις διαπραγματεύσεις του TTIP πρέπει να βγει το οπτικοακουστικό, ο οπτικοακουστικός τομέας. Ε, Δυστυχώς όμως δεν μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε αυτή την ε, πλήρη εξαίρεση και έχουν μείνει ορισμένα παραθυράκια ανοιχτά που θα δώσουν τη δυνατότητα να ξαναμπεί το θέμα αυτό, το τομέα αυτό στις διαπραγματεύσεις. Ε, ξέρετε ότι πολλές φορές έχουμε προσπαθήσει εμείς με τις, ε, με, στα διάφορα διαπραγματευτικά επίπεδα πόσο μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτήν την εξαίρεση διότι στα από τα οπτικοακουστικά υπάρχει εξαίρεση των υπηρεσιών αλλά όχι των επενδύσεων. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και αν έχω ερμηνεύσει σωστά ε, τα λεξέντα ε, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της Ιταλικής Προεδρίας αλλά και πέραν της Ιταλικής Προεδρίας θα προσέξετε ιδιαίτερα και θα παρακολουθείτε ιδιαίτερα τις εξελίξεις έτσι ώστε να μην θυσιαστούν τα οπτικοακουστικά μέσα στο βωμό του TTIP. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα και χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω ότι η Ιταλική κυβέρνηση είναι στο πλευρό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχω μία ερώτηση ε, στον Υπουργό Οπτικοακουστικών και Ψηφιακών Μέσων. Είπατε ότι και στο, θα ασχοληθεί η Ιταλική Προεδρία με αυτό το θέμα και αναγκαστικά ε, θα συμμετάσχει και στον τριμερή διάλογο για τα ψηφιακά μέσα. Είναι ένα εμπεριστατωμένο ντοσιέ αυτό, αλλά ιδιαίτερα πρόσφατα υπήρχε μεγάλη αντίδραση έναντι των σχεδίων της Κομισιόν και με μεγάλη πλειοψηφία το σώμα δήλωσε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να διατηρηθεί η ουδετερότητα Υπάρχουν ορισμένες υπηρεσίες που μπορούν να διακυβεύσουν την ουδετερότητα. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ σαφείς και αυστηροί και έχουμε υποβάλει και συγκεκριμένες προτάσεις. Από ό,τι ξέρουμε οι διαπραγματεύσει στο Συμβούλιο είναι πολύ δύσκολο, διότι υπάρχουν ε, διαφορετικές απόψεις και στο επίπεδο των κυβερνήσεων. Γι' αυτό λοιπόν ε, το ερώτημα είναι θα σταθείτε στο πλευρό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο θέμα των ψηφιακών μέσων και ε, η δική μας στάση που πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ισορροπημένη και εξασφαλίζει και την ουδετερότητα. Είναι πολύ σωστή λοιπόν, διότι χρειαζόμαστε μια ουδετερότητα για την πολιτισμική πολυπλοκο... Ε, πολιτισμικότητα, πολυπολιτισμικότητα ε, για την διασφάλιση των, των διαφορών και των πολλών πολιτιστικών εκδηλώσεων, το οποίο σίγουρα προωθείται μέσω των ψηφιακών μέσων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λιμπάτσκα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε, ευχαριστώ πολύ για τις εισηγήσεις σας κύριε Υπουργή ε, που παρουσιάσατε ακριβώς τις προτεραιότητες της Ιταλικής ε, Προεδρίας. Δύο θέματα θα ήθελα να θίξω ε, τα οποία αναφέρατε, τα οποία ανέφερε ο κύριος θα ήθελα να ε, συμφωνήσω μαζί σας ότι η Ευρώπη πρέπει να ανακτήσει χαμένο έδαφος έναντι του υπόλοιπου κόσμου. Όμως, σε έναν τομέα είμαστε ηγέτες, ηγούμεθα, είμαστε ε, πρωτοπόροι στον πολιτισμό, στα πολιτιστικά θέματα, ας το πούμε κουλτούρα στο, αναφέρεται και το πρόγραμμα Εράσμους ή τη νέα μορφή την οποία θα έχει το Εράσμους και όπως είπατε ε, η ψηφιακή επανάσταση ε, πρέπει οπωσδήποτε να, να βασίζεται και στα πνευματικά δικαιώματα. Ε, πιστεύω ότι αυτή η επανάσταση θα θα, φέρει, θα επιφέρει πολλά ωφέλη και δεν θα δημιουργήσει προβλήματα και ζημίες, διότι οι νέοι άνθρωποι θέλουν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους ε, και τα συναισθήματά τους αυτά μπορούν να τα εκφράσουν όταν έρχονται σε άμεση επαφή με πολιτιστική και από πολιτιστικές εκδηλώσεις. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε την πολιτιστική έκφραση, την ελευθερία της έκφρασης και να ε, προωθήσουμε τους νέους ε, στην κατανάλωση πολιτιστικών προϊόντων έτσι ώστε όχι μόνο να υποφελούνται από το διαδίκτυο, το ίντερνετ και τα ψηφιακά μέσα αλλά και από όλα τα άλλα προγράμματα που είναι στη διάθεσή τους. Το πρόγραμμα Εράσμους λοιπόν θα πρέπει στις προτεραιότητες του να δίνει τη δυνατότητα στους νέους να έρθουν σε άμεση επαφή με τον πολιτισμό, με πολιτιστικούς τομείς και να διευκολύνει την άμεση ε, επαφή τους με την τέχνη. Και γι' αυτό θα πρέπει ιδιαίτερα να, διασφαλίσουμε και να προωθήσουμε την πρόσβαση στο διαδίκτυο και στα ψηφιακά μέσα. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Κύριε, κύριε Η κυρία Νίβολ Αντινόλφη, ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι προτάσει τη Ιταλική Προεδρία είναι καλά λόγια βεβαίω και θα θέλαμε να καταλάβουμε ωστόσο τι θα κάνει η Προεδρία στην πράξη, λαμβάνοντα υπόψη ότι παρουσιάζει ένα πρόγραμμα τώρα μόνο όταν έχει περάσει σχεδόν το 1 τρίτο του εξαμήνου. Είναι γεγονό ότι σε πολλέ περιπτώσει η πολιτιστική κληρονομιά είναι δυσπρόσιτη. Πώ θα αντιμετωπίσει τα θέματα που το ψήφισμα του ΙΕ για τα δικαιώματα των ε, αναπήρων στην πολιτιστική κληρονομιά, πώς θα υλοποιήσει την ανάδειξη των ε, άειλων ε, πολιτισμικών αγαθών της Ευρώπης, τι θα κάνει για τα ίσονο σημασία πολιτιστικής κληρονομιάς, γιατί συχνά τα κονδύλια πηγαίνουν στα μεγάλα ελκυστικά ε, ε, εργαλεία τουρισμού που χρησιμοποιούνται στην ουσία μόνο για την προσέλκυση τουριστών. Πόσο ο Υπουργός ε, θα βοηθήσει τον, δημιουργικό, τον κόσμο των δημιουργών, μήπως θα μπορούσε να γνωρίζουν περισσότερο οι Ευρωπαίοι τον διαγωνισμό που εσείς αναφέρατε, ε, την δυνατότητα δηλαδή να χρησιμοποιούνται ε, να χρησιμοποιούνται ε, δραστηριότητες της, των δημιουργών μόνο και μόνο χωρίς καμία αποζημίωση. Και τέλος, το πώς θέλει να, να προωθήσει η Προεδρία την ανάδειξη των, όλων των πολιτιστικών αγαθών. Θα προτείνει και εδώ τις ε, συμφωνίες ιδιωτών και δημοσίου όπως αυτή που κάνετε στη Ρόνη με την εταιρεία αυτοκίνητων δρόμων για τη διαχείριση της, ε, ενός από τους παλαιότερους δρόμους του κόσμου την, ε, την Άπη Αντίκα. Μήπως θα έπρεπε να προωθήσετε αντί των επιχειρήσεων τους, τους διαχειριστές του πολιτισμού και τους γνώστες των θεμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μαλτέζε. Στα ευρωπαϊκά θέματα να μείνετε αν γίνεται, που είναι αντικείμενο της συζήτησης σήμερα. Κύριε Υπουργέ, προσπαθείτε εδώ και καιρό να αναδείξετε την οικονομική σημασία του πολιτισμού και να αναφέρεται ότι ο πολιτισμός θα μπορούσε να είναι ένας από τους βασικούς ε, τομείς όπου μπορεί να βρεθεί λύση για την τραγωδία της ανεργίας των νέων. Εγώ συμφωνώ με την θέση σας. Υπάρχει ωστόσο ένα πρόβλημα προστασίας της, των υφιστάμενων θέσεων εργασίας. Όπως ξέρετε, ε, εγώ μπήκα πολύ νέος ε, στον, στην αγορά εργασία. Αν συγκρίνω την εποχή που μπήκα εγώ στη δημοσιογραφία με έναν ε, νέο δημοσιογράφο, ίσως και μεγαλύτερο από μένα, εγώ μπήκα 18, αυτός ας πούμε είναι τριαντάρης, και εδώ τον μισθό του τριαντάρη δημοσιογράφου σήμερα, τι ποιότητα πιστεύετε ότι θα έχει η ενημέρωση που είναι ένας από τους πυλώνες της δημοκρατίας μας. Το ίδιο ρωτώ όταν κοιτώ τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων ε, στα θεάματα. Ε, δεν είναι μόνο το πρόβλημα η απειλή των συγγραφικών δικαιωμάτων, αλλά το ότι η αγορά της, ε, η πολιτισμική αγορά χάνει την σταθερότητα των θέσεων των εργαζομένων σε αυτόν. Πώς μπορεί η Ιταλική Προεδρία να εξασφαλίσει στην Ευρώπη μεγαλύτερη προστασία και καλύτερους μισθούς για τους εργαζόμενους στον κλάδο του πολιτισμού. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Διακόνου. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, ένα σπίτι από την αρχαία Ρώμη είπε και νομίζω ότι είχε δίκιο ότι κάθε καλλιτέχνης πρέπει να είναι δυστυχής. Και όντας δυστυχής Πιστεύω ότι η δυστυχία του σημερινού καλλιτέχνη είναι υποχρεωτική. Όμως, παρόλα αυτά, ανησυχώ που θα οδηγήσει αυτή η δυστυχία. Δηλαδή, έχει αρχίσει να μετατρέπεται σε μια πολιτιστική κληρονομιά αυτή η δυστυχία. Γι' αυτό ανησυχώ. Πριν από δύο λεπτά μου είπαν ότι θα είμαι εισηγητής για την πολιτιστική κληρονομιά και είμαι ευτυχής γι' αυτό. Αυτό σημαίνει ότι αν και πρόκειται να σας ε, υποβάλω μια ερώτηση, τελικά δεν θα σας την υποβάλω, διότι οι απαντήσεις σας υπήρξαν σαφείς σήμερα το απόγευμα. Μας δώσατε καλά νέα, ιδιαίτερα για την πολιτιστική εξαίρεση. Προέρχομαι από τη Ρουμανία και είχαμε μια τραγική εμπειρία απαγορεύσεων για δεκαετίες Τώρα πια που δεν είμαστε κάτω από τον κομμουνισμό, μπορώ να σας πω ότι οι οικονομικές απαγορεύσεις είναι αυτές που είναι φοβερές και εξαντλητικές. Και αν δεν μπορέσουμε να υπερασπίσουμε τους εαυτούς μας, θα εξαφανιστούμε. Και όπως είπε ο υφυπουργό, σωστά, θα πρέπει να μιλάμε όλες τις γλώσσες και όχι μόνο μία σε αυτή την επικράτεια, την ευρωπαϊκή οι Αμερικανοί φίλοι μας έχουν ένα κόμπλεξ σε σχέση με την Ευρώπη που αφορά τον πολιτισμό της. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας αυτό και να προασπίσουμε τους εαυτούς μας. Και γι' αυτό επιμένω ότι πρέπει να συνεργαστούμε όλοι σε αυτού τους τομείς. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για τις καλές σας προθέσεις και ελπίζω να ξανασυναντηθούμε. Ευχαριστώ. Ε, grazie onorevole Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε και κύριοι Υπουργοί. δεν θα πρέπει να δούμε την, τον πολιτισμό και την τέχνη από την πλευρά της, ε, από τη σκοπιά της εμπορικής ε, πολιτικής. Εδώ θέλουμε να υποστηρίξουμε την πολυπολιτισμικότητα ε, και την παιδεία και επιμόρφωση των νέων. Γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω Ποιο είναι το πρόγραμμα της Ιταλικής Προεδρίας για την κατάρτιση των νέων και τι κονδύλια θα διαθέσει. Η Πρόεδρος. Έχουμε ακόμα δύο συναδέλφους πριν δώσω το λόγο. Γκέρμανς Μίτσι, ο κ. Εύανς πρώτα και μετά οι άλλοι δύο συνάδελφοι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους υπουργούς για την παρουσίαση που μας έκανα. Συμφωνώ και εγώ με την πολιτιστική εξαίρεση. Είπατε κι εσείς ότι ο πολιτισμός είναι υπερβολικά αξιόλογος και πολύτιμος για να μην χρησιμοποιηθεί, τον διαχειριστούμε διαφορετικά. Μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα θέματα με την νεολαία. Ένα πρόγραμμα παρόμοιο με το Εράσμους, αλλά περισσότερο πόλης πολυπολιτιστικό και η αδελφοποίηση μουσείων και μνημείων είναι μια καλή ιδέα. Εκπροσωπώ την Ουαλία στο Ευρωκοινοβούλιο, στο Ευρωκοινοβούλιο και όλα αυτά είναι σημαντικά για μας. Ο πολιτισμικός τουρισμός αφήνει πάνω από 50 εκατομμύρια την ημέρα στην οικονομία μας και μας ενδιαφέρουν οι εταιρικέ σχέσεις με άλλες χώρες αλλά είμαστε μια μικρή δίγλωση χώρα, ε, τα ουαλικά δεν είναι επίσημα γλώσσα αλλά ελπίζω ότι στο πρόγραμμά σας θα περιλαμβάνουμε και τις ε, γλώσσες των μειονοτήτων που δεν είναι επίσημα αναγνωρισμένες, διότι παίζουν σημαντικό ρόλο στο διαδίκτυο και στα μίδια. Πρέπει να τις περιλάβουμε αυτές τις ε, γλώσσες για να, ε, για να περιλάβουμε όλοι το, τον πολιτισμό της Ευρώπης. Συνάδελφος Μίτση, σας ευχαριστώ, ευχαριστώ τους υπουργούς Λυπάμαι που παρατηρώ ότι περισσότεροι από τους συνάδελφους μου μιλούν στην ε, μητρική τους γλώσσα. Και σε αυτή την επιτροπή που είναι τόσο σημαντικός ο πολιτισμός και η πολυπολιτισμικότητα, λυπάμαι που τα μαλτέζικα που είναι επίσημη γλώσσα α, της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει διερμηνία. Θα μιλήσω λοιπόν αγγλικά υποχρεωτικά. Υπουργοί, Ε, κατάλαβα τη βασική προσέγγιση της ομιλίας σας και τη σπουδαιότητα που αποδίδεται στον πολιτισμό και στην παιδεία. Ε, η Ιταλική Προεδρία είναι καλό νέο. Ε, θα ψηφίσουμε αύριο για τον προϋπολογισμό. Και ο προϋπολογισμός αύριο έχει υπογραμμίσει τη δημιουργικότητα της Ευρώπης, την Ευρώπη των πολιτών και ασχολείται και με το Erasmus Plus. Οι συνάδελφοι μίλησαν για το πόσο σημαντική είναι η παιδεία, η μαθητεία, η κατάρτιση. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για τα παιδιά μας, τους νέους μας, για να έχουν ένα καλό μέλλον. Όλοι ξέρουμε λοιπόν τη σπουδαιότητα της παιδείας και τη διασύνδεσή της με την εργασία. Τώρα, δυστυχώς η Κομισιόν έχει προτείνει μια πολύ μικρή αύξηση του κονδυλίου για την παιδεία. Ενώ οι ευρωβουλευτές ζητούν αύξηση. Το ερώτημα μου προς εσάς λοιπόν είναι, η Προεδρία τι θα υποστηρίξει, την αύξηση του προϋπολογισμού ή όχι. Θέλουμε λοιπόν να υποστηρίξετε την αύξηση του, προ... του κονδυλίου για την παιδεία, γιατί είναι πολύ σημαντικό για την νεολαία μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για την συμμετοχή τους και τα ερωτήματα που έθεσαν. Πριν δώσω το λόγο στους εκπροσώπους του, της Ιταλικής Προεδρίας ε, να απαντήσω στην ερώτηση για τη γλώσσα. Έχουμε κάποιες ε, ελλείψεις σε γλώσσες, τα Μαλτέζικα για παράδειγμα, λόγω του ότι και η αίθουσα που έχουμε είναι μικρή, δεν έχει μεγάλο αριθμό ε, από καμπίνες και δεν έχουμε και αρκετούς διερμηνείς. Δίνω το λόγο στους δύο υπουργούς με δύο θέματα. Πρώτον, ακούσατε κύριε Υπουργή πόσο η Επιτροπή μπορεί να είναι σύμμαχος, φυσικός σύμμαχος του σύμμαχό σας στο Συμβούλιο του Υπουργών εάν προωθήσετε τις προτάσεις που θέσατε τώρα ως προτεραιότητα και που συμμεριζόμαστε εμπολείς και εμείς την οριζόντια, εγκάρσια, ε, συμπεριληπτική προσέγγιση του πολιτισμού στις πολιτικές της Ένωσης. Για το λόγο αυτό θα έχουμε και συνάντηση με τους συντονιστές των ομάδων προφανώς, αλλά θέλω να πω ότι ως πρόεδρος της Επιτροπής, προσωπικά δηλαδή, να σας πω ότι μια ευχή που θα μπορούσαμε να απευθύνουμε προς την Ιταλική Προεδρία είναι ότι θα θέλαμε και ο νέος Επίτροπος στον πολιτισμό να έχει, που έχει, να έχει σοβαρά, σοβαρό χαρτοφυλάκιο, ε, να μην μειωθούν οι αρμοδιότητες του και ό,τι έχει να κάνει με το περιεχόμενο online, οπτικοκουστικό και ψηφιακό, να είναι αρμοδιότητα του, του Επιτρόπου Πολιτισμού, ανεξάρτητα από τις Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής. Το λέω για τους νέους συναδέλφους αυτή τη στιγμή. Οι Γενικές Διευθύνσεις Πολιτισμού, Connect, εσωτερικής αγοράς και όχι διεθνούς αγοράς, συχνά ε, διασπείρουν τις αρμοδιότητες της Επιτροπής στον τομέα του πολιτισμού. Θα ήθελα, θα ήλπιζα ο νέος Επίτροπος Πολιτισμού να έχει μεγαλύτερη παρουσία και πιο ισότιμη θέση, ούτως ώστε να μπορεί να χρησιμοποιεί πλήρως τη θέση του, κάτι που το που το ανέφερε και ο κ. Τζακομέλα και ο κ. Φραντσεσκίν για το θέμα του copyright να μπορεί να έχει ε, πολύ σοβαρή παρουσία. Δίνω το λόγο στον Υπουργό για να απαντήσει. Σύντομα, πολλές παρεμβάσεις, σας χρήσιμες, ευχαριστώ. Δείχνουν και κοινή, κοινά συναισθήματα, κοινές ευαισθησίες προτάσεις ήταν περισσότερο παρά ερωτήματα ενδεχομένως για την πολιτιστική εξαίρεση. Προφανώς θα υποστηρίξω την αρχή αυτή και πέραν της τελικής προεδρίας. Πιστεύω ότι η αρχή αυτή πρέπει να εξηγηθεί καλά και να βρούμε μια κοινή σύνθεση για να αποφύγουμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον τα ίδια προβλήματα. Αυτό το θέμα θα συζητηθεί και στην επίσημη συνάντηση των Υπουργών το Δεκέμβριο. Θα ήταν αντιπαραγωγικό να δημιουργηθούν μέτωπα χωρών μέσα στην Ένωση που παρετίθενται μεταξύ τους. Καλύτερο είναι να χρησιμοποιήσουμε, ε, να φτιάξουμε μια κοινή θέση με υπογραμμίζοντας το ότι δεν μιλάμε για πολιτικές προστατευτισμού, αλλά για να εξηγήσουμε ότι προς το παρόν πρέπει να αφαιρέσουμε τον κλάδο του πολιτισμού από τα εμπόδια. Εδώ περιλαμβάνουμε τα οπτικοακουστικά, τον κινηματογράφο. Να μην υπαχθούν δηλαδή αυτά στην απλή... Ε, να μην υπαχθούν και να μην υποταχθούν στην απλή λογική της αγοράς. Ένα καλό βιβλίο βέβαια είναι καλό βιβλίο ακόμα και αν δεν πουλιέται. Η αγορά δεν μπορεί να είναι το μόνο σημείο αναφοράς. Πρέπει να είναι ένα σημείο αναφοράς, αλλά όχι το μόνο σημείο αναφοράς της ε, πολιτιστικής δραστηριότητας. Θα πρέπει να μπορούμε να εξηγήσουμε στους συνομιλητές μας και στην τελευταία συνάντηση η Επιτροπή δεσμεύτηκε να ακολουθήσει την θέση αυτή για την πολιτιστική κληρονομιά να εξηγήσει ότι δεν είναι ένα θέμα εμείς, δηλαδή το ζήτημα δεν είναι μια αντιπαράθεση μεταξύ ημών και των εταίρων μας, αλλά ένα κοινό θέμα. Μίλησα για το Εράσμους. Χρησιμοποίησα το Εράσμους για να γίνω κατανοητός. Το Εράσμους αφορά την εκπαιδευτική περίοδο. Εγώ μιλούσα για κάτι που ξεπερνά την περίοδο της εκπαίδευσης. Ανταλλαγή καλλιτεχνών, ανταλλαγή πολιτιστικών εμπειριών. Θα ήθελα ένας νέος που δούλεψε σε ένα μεγάλο μουσείο στη χώρα μου να έχει μια εμπειρία σε ένα μουσείο μιας άλλης χώρας. Ένας βιβλιοθηκάριος, ένας αρχιοθέτη σε μια ευρωπαϊκή χώρα να μπορεί να βοηθηθεί για να πάει σε μια άλλη χώρα να δουλέψει εκεί. Αυτό θα επιτρέπε, θα λειτουργεί με υπόδειγμα την χρηματοδότηση του Εράσμους, αλλά που θα ε, επιτρέπουν την ανταλλαγή νέων καλλιτεχνών, δημιουργώντας κοινή ηθαγένεια, κοινή συνέργεια. Να απαντήσω στην κυρία Τινόρη ότι δεν απαντώ σε ιταλικά εσωτερικά πολιτικά ζητήματα, αλλά να σας πω ότι ο διαγωνισμός που αναφέρεται προέβλεπε τη δυνατότητα και δεν δημιουργήθηκε φέτος, ήταν και τα προηγούμενα έτη, προέβλεπε τη δυνατότητα επίσκεψη, τέλος πάντων να πας σε μεγάλα, να στείλει ε, ε, σε μεγάλα μουσεία ε, δωρεάν νέους. Το να παίξει στην πινακοτέκα της Μπρέρα ένας νέος δεν είναι κάτι, κάτι αμεληταίο. Εγώ θεώρησα ότι το να στέλνουμε νέους καλλιτέχνες στο τζάπα δεν έδινε το σωστό μήνυμα και το κατήργησε. Το θέμα ωστόσο αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να συμπεριλάβει, να, να εξετάσει το θέμα της προστασίας της πολιτικής κληρονομιάς ευρύτερα και χωρίς ταμπού. Δεν θέλουμε να πούμε ότι ε, θα εγκαταλείψουμε το ρόλο του δημοσίου τομέα στην προστασία της πολιτιστική κοινωνίας, ότι αυτό θα μείνει στα χέρια των ιδιωτών. Ούτε, αλλά γιατί να αρνηθούμε μορφές συνεργασίας ή οικονομικής συνεισφοράς των ιδιωτών για την ανάδειξη ή την προστασία των πολιτιστικών προϊόντων. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κρατήσουμε ανοιχτό. Επιπλέον, η προστατευμένες περιοχές της UNESCO ε, ονομάζονται πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας. Άρα το αγαθό αυτό είτε ανήκει σε έναν ιδιώτη είτε σε ένα κράτος ε, έχει κάποιον μεταβατικό χαρακτήρα. Όλοι είμαστε μεταβατικοί. Η, ανθρωπότητα κερδίζει από αυτή την πολιτιστική κληρονομιά. Για τον κύριο Μαλτέζε, το θέμα της ε, Επισφάλεια των θέσεων εργασίας στον τομέα του πολιτισμού δεν είναι μόνο θέμα του τομέα του πολιτισμού. Θα ήθελα να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας στον ε, τομέα. Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τον πολιτισμό για την ανάδειξη της κληρονομιάς, θα έπρεπε να το κάνουμε δημιουργώντας σταθερότερες θέσεις εργασίας, λιγότερο επισφαλής αλλά και περισσότερες και το λέω διότι, ε, ε, ξέρετε, η ιδέα της ευτυχίας του καλλιτέχνη είναι ένα ρομαντικό στοιχείο. Μπορεί ωστόσο κάποιος να έχει εξαιρετική ποιότητα, έστω και αν ε, ιδίως αν η ευτυχία τον βοηθά, όχι μόνο όταν είναι δυστυχής. Η ιστική πολυμορφία που πρέπει να προστατεύσουμε δεν έχει μόνο τουριστική διάσταση. Η ποικιλομορφία, η πολιτιστική ποικιλομορφία είναι ο πλούτος μας. Μπορεί να γίνει στοιχείο δύναμης, όχι αδυναμίας. Και ρωτήθηκε πώς γίνεται η χρηματοδότηση. Ε, αυτό είναι ένα θέμα. Η δημιουργική Ευρώπη ε, μεταξύ των στόχων της έχει και την προώθηση και διαφύλαξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Υπάρχει λοιπόν το εργαλείο αλλά όπως και άλλα πράγματα ε, αναφέρθηκαν, υπάρχουν τα εργαλεία, οι πόροι λείπουν. Η τελευταία παρέμβαση με, με ρώτησε τι θα κάνουμε μετά. Ισορροπία πρέπει να κρατήσουμε για το θέμα των προϋπολογισμών. Η μείωση είναι σημαντικό, αλλά αυτό προκύπτει από τις θέσεις των ε, κρατών. Η Προεδρία πρέπει να διαμεσολαβήσει μεταξύ των κρατών, αλλά πρέπει να σεβαστεί τις αποφάσεις. Αν με, ρωτήσετε ποια είναι η θέση μου ως Ιταλού, θα σας έλεγα ότι και τώρα και στο μέλλον είμαι υπέρ της ε, ε προστασίας του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ελπίζω αυτό να είναι ένα επιχείρημα που θα περάσει στο Συμβούλιο. Θέλετε να απαντήσετε, κύριε Τζακομέλη, ε, για τα θέματα της δικής σας αρμοδιότητας. Μπορώ να δώσω. Καταρχάς, σας ευχαριστώ. Ε, να απαντήσω στην κυρία Καμερέβερτ. για την πρόσταση της Προεδρίας ό,τι αφορά το net neutrality. Ειδικότερα την θέση του Κοινοβουλίου και ενισχύοντας περαιτέρω τις θέσεις της κυρίας Κρούζ και το αν συμμεριζόμαστε ή όχι. Εμείς συμφωνούμε απόλυτα με την αρχή της ε, ουδετερότητας του διαδικτύου. Το συζητήσαμε χτες στην Επιτροπή που ασχολείται με το θέμα. Στους ε, τριλόγους θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με ειλικρίνεια το θέμα. Αν κατάλαβα καλά τη θέση του Κοινοβουλίου και το πνεύμα που το εμπνέει είναι ότι η ουδετερότητα του δικτύου εξασφαλίζει ότι το δίκτυο είναι ενιαίο, ελεύθερο, ανοιχτό, εκμεταλλεύσιμο, χώρος ευκαιριών, χωρίς επικάλυψη ή μικρότερη με μεγαλύτερη ταχύτητα να με το ποιο πληρώνει και πόσο. Εμείς πιστεύουμε για τις εξειδικευμένες υπηρεσίες πρέπει να παρασχεθεί δυνατότητα ανάπτυξης που δεν θα οδηγεί στο να δημιουργεί de facto ίντερνετ πολλών ταχυτήτων μεταξύ αυτών που πληρώνουν υπηρεσίες και αυτών που δεν πληρώνουν. Άρα δεν ξέρω αν ο όρος που χρησιμοποιήθηκε περιορισμός των υπηρεσιών είναι σωστός ή όχι, είναι να επιτρέψουμε μια ανάπτυξη που δεν θα υπονομεύει την αρχή της ε, ουδετερότητας. Το θέμα είναι ότι αυτό δεν μπορεί να οδηγήσει στην, στο λιγοπόλιο κάποιων μεγάλων ομίλων που αποφασίζει στην πράξη ποια θα είναι, ποια, ποιος πολιτισμός θα εκφράζεται, ποια φωνή θα ακούγεται, ποιο μήνυμα θα περνάει στον πολίτη. Το ανοιχτό δίκτυο σημαίνει ανοιχτό πραγματικά χώρο ευκαιριών και φοβάμαι ότι η συζήτηση σήμερα είναι λίγο πιο δεσμευτική από αυτή που το Κοινοβούλιο και, το, και η Επιτροπή είχαν εξετάσει στο παρελθόν. Σας είπα ότι στις Ηνωμένε Πολιτείες προσπάθησαν να, να κάνουν μια συμφωνία με τα Telecom, με τις τηλεπικοινωνίες. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι θα υπάρξει συμφωνία των μεγάλων επιχειρήσεων για το τι πρέπει να για το πώς πρέπει να, να, πληρώνεται η χρήση του ε, φάσματος. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι τα παιδιά που σε ένα ε, γκαράζ δημιουργούν μια εφαρμογή που επιτρέπουν να γεννηθεί ένα μεγάλο πολιτιστικό και ε, οικονομικό γεγονός θα είναι αντικείμενο μύθου, δεν θα είναι πραγματικότητα. Αυτός δηλαδή μόνο που θα έχει στις πλάτες του χρήματα θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο. Εμείς πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να αποφευθεί κάτι τέτοιο. Γι' αυτό προτείνουμε στις κυβερνήσεις της Ευρώπης να προσπαθήσουμε από κοινού τους ώστε να μην συμβεί κάτι τέτοιο και να επιτρέψουμε σε όλους την δίκαιο, τον δίκαιο ανταγωνισμό και να φροντίσουμε το ώστε το διαδίκτυο θα παραμείνει χώρος ευκαιριών για όλους ανεξάρτητα από την οικονομική ικανότητα που έχει από πίσω του. Ευχαριστούμε και για τη διαφάνεια, την σαφήνεια συγγνώμη που αναφέρεται και εμείς ε, είναι ένα θέμα που πρέπει να ε, επεξεργαστούμε. Ευχαριστώντας κλείνω, κλείνω ευχαριστώντας τους δύο υπουργούς, ε, ο κ. Τζακομέλη, να θυμίσω ότι θα γίνει στις 24 Οκτωβρίου στη Ρώμη μια διάσκεψη για τα οπτικοακουστικά, ακριβώς για το θέμα της αγοράς και της διαχείρισης των οπτικοακουστικών. Πιστεύω ότι θα είναι και μια ευκαιρία για όποιον θέλει να συζητήσει το θέμα. Σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία και Ελπίζω να είσαστε συνεκτικοί και σε αυτά που είπατε για τον προπολογισμό. Έχετε τώρα ο κύριος Μπόμπα για τις Ιταλικές προτεραιότητες ε, για τον αθλητισμό και την πολιτική των νέων.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

Έρχεται ο κύριος Μπόμπα. Καθίστε συνάδελφοι. Καλωσορίζω τον κύριο Μπόμπα. Συνάδελφοι, έχουμε και συνάντηση των συντονιστών, οπότε πρέπει να τελειώσουμε γρήγορα. Allora, eh, Καθίστε και μην μιλάτε αν γίνεται. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας. Η ησυχία. Έχω λέω τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Λουίτζι Μπόμπα, υφυπουργό εργασίας και κοινωνικών πολιτικών με έμφαση, με αρμοδιότητα για τις πολιτικές νέων. Να μου τονίσω ότι είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα μου, διότι αυτό σημαίνει ότι η εγγύηση για τους νέους, η πολιτική δηλαδή και η πολιτική που υπάρχει στο Εράσμος περιλαμβάνονται σε, μια, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο των πολιτικών προνοίας. Παρακαλώ τον κύριο Μπόμπα να μας παρουσιάσει μαζί με τον κύριο Πανεμπιάνκο που είναι ειδικό ε, για το θέμα πολιτικής ε, αθλητισμού. Η, η εκπροσώπηση αφορά άλλο Υπουργείο. Ζητώ καταρχάς να μιλήσουμε για πολιτικές νέων και μετά τα θέματα της πολιτικής αθλητισμού. Ο κύριος Μπόμπα. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Οι δύο τμήματα θα έχει ομιλία μου. Πρώτον, πολιτικές για τους νέους. Δεύτερον, πολιτικές για τον αθλητισμό. γιατί ο υφυπουργό Δεδίο δεν μπορούσε να έρθει, που είναι αρμόδιος, έχει σήμερα Υπουργικό Συμβούλιο στην Ιταλία. Πρώτον, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έχουν από καιρό θέση τις πολιτικές για τους νέους ως βασικό στοιχείο και για τη μάχη κατά της ενεργείας και ως τρόπο ανανέωσης του κοινωνικού και οικονομικού μοντέλου της Υπήρου. Όλα αυτά με επίγνωση ότι οι νέοι αποτελούν, αντιπροσωπεύουν ένα παράδοξο. Αφενός καλούνται να ενταχθούν στην κοινωνική και ε, οικονομική ζωή, αλλά ταυτόχρονα είναι και δυνάμεις καινοτομίας και, και αλλαγής. Άρα ε, ε, ενσαρκώνουν τις μελλοντικές δυνατότητες. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ωστόσο ότι η στρατηγική της Ένωσης για τους νέους του 2010, για την περίοδο 2010-2018 που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 27 Νοεμβρίου του 2000, ε, στις 17 Νοεμβρίου του 2009 στηρίζεται σε δύο βασικούς άξονες. Πρώτον, τη δημιουργία ευκαιριών για τους νέους μέσω της εκπαίδευσης και της ένταξης της εργασίας και δεύτερον την προώθηση μιας ενεργού ηθαγένειας και κοινωνικής και ουσιαστικής ε, κοινωνικής ένταξης. Η στρατηγική αυτή ε, συνδέει πολύ καλά το διώνυμο νέοι ικανότητες. Οι ικανότητες που αποκτούνται και στην τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση, αλλά και άτυπη που με στόχο την επίτευξη ενός πραγματικού ευρωπαϊκού διαβατηρίου δεξιοτήτων. Η Ιταλία στην προεδρία της προτίθεται να προωθήσει εκ νέου μια ενοποιημένη, ολοκληρωμένη προσέγγιση των πολιτικών για τους νέους που θα αντιμετωπεί, που θα κάνει τον εγκάσιο χαρακτήρα των πολιτικών αυτών ως κεντρικό στοιχείο γιατί θα προσανατολίζεται και στην ανάπτυξη της αυτονομίας των νόμων και στην υποστήριξη των δυνατοτήτων να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την ε, ε, βελτίωση των συνθήκων τους. Δυστυχώς, ωστόσο, η αυτονομία αυτή τίθεται σε κίνδυνο από πολλούς παράγοντε που η κρίση που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια ε, ε, όξινε περαιτέρω. Δεν είναι τυχαίο στην τελευταία έκθεση για τους νέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρθηκε ότι οι νέοι παραμένουν η πιο εκτεθειμένη κοινωνική ομάδα και σε φαινόμενα αποκλεισμού και σε φαινόμενα φτώχειας, αλλά και στην, και στην ένταξη σε κακοπληρωμένες ή επισφαλείς θέσεις εργασίας. Ο στόχος της Ένωσης είναι να υπάρξει πλήρης εκμετάλλευση των δικαιωμάτων από τους νέους, όχι μόνο να υπάρχουν τα δικαιώματα όνομα ταυτόχρονα να προωθήσει το πέρασμα από την εξάρτηση των νέων στην αλληλεξάρτηση. Το Συμβούλιο των Υπουργών για την ε, Παιδεία και την Νεολαία σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα πλάνο εργασία για το 2014-2015 επέλεξε το τρίο της Προεδρίας Ιταλία, Λετωνία, Λουξεμβούργο με το θέμα του empowerment. Η Ιταλική Προεδρία στο πλαίσιο αυτό επέλεξε να ασχοληθεί περισσότερο με την προώθηση στην πρόσβαση των δικαιωμάτων, ούτω ώστε να ενθαρρύνει την αυτονομία των νέων και την, συμμετοχή, την κοινωνική συμμετοχή τους. Προς, αυτή, ε, προς το σκοπό αυτό στάληκε ένα κείμενο σε όλα τα κράτη-μέλη. Επίσης η Προεδρία θέλησε να δώσει έμφαση στα θέματα της πολιτικής απασχόλησης, υποστηρίζοντας την απασχόληση των νέων, ενθαρρύνοντας την κινητικότητα και εργασιακή και κοινωνική και καθιστώντας την αγορά εργασίας πιο συμπεριληπτική. Ε, είναι σημαντικό ότι σε όλες τις χώρες ε, προχωρά το πρόγραμμα εγγύησης νέων. Τέλος, η Προεδρία θέλει να αξιοποιήσει ιδιαίτερα το, την πολιστική κληρονομιά και τις διαφορετικότητες του πολιτισμού αλλά και την ικανότητα των νέων να ενταχθούν σε δημιουργικές διαστάσεις ως εργαλείο που είναι σημαντικό και εν ώψη του νέου προγράμματος εργασίας του Συμβουλίου για τον πολιτισμό από το 2015 έως 2018. Στο πλαίσιο αυτό του γενικού ορίζοντα των πολιτικών της Προεδρίας Θέλω να αναφερθώ στο θέμα της εκμάθησης των δεξιοτήτων κλειδιών προς δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, μια δράση προς τους νέους στον τομέα της εμβάθυνσης, της εκμάθησης, της άτυπης εκμάθησης, ε, συμμετοχή, εθελουσία, συμμετοχή σε κοινωνικές οικονομικες δράσεις και δεύτερον, δράσεις ένταξης που στηρίζονται, όπως έλεγα, σε μια εγκάρσια προσέγγιση σε κάθε τομέα που επηρεάζει τη ζωή των νέων. Επαναλαμβάνω, η εγκαρσιότητα είναι βασικό εργαλείο για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών για τους νέους. Τα συμπεράσματα στα οποία θα πρέπει να φτάσει το Συμβούλιο θα στηριχθούν σε τρία θέματα ικανότητα άσκησης της πρόσβασης στα δικαιώματα, δουλειά, πίστη, σπίτι, να ενθαρρύνουμε την, κοινωνικο-εκπαιδευτική ε, ανάδειξη και να υπάρξουν διατομεακές παρεμβάσεις που θα είναι στο κέντρο μιας ευρωπαϊκής διάσκεψης για την νεολαία που θα γίνει στη Ρώμη από τις 13 μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. Ο στόχος της διάσκεψης είναι ένα κοινό έγγραφο για την πρόσβαση στα δικαιώματα. Το κείμενο αυτό με τη σειρά του θα τροφοδοτήσει την πρόταση συμπερασμάτων του Συμβουλίου που θα γίνει στις 12 Δεκεμβρίου του 2014. Το Συμβούλιο πριν το Συμβούλιο θα γίνει ένα γεύμα εργασία που θα έχει στόχο να καταλήξουμε συμπεράσματα για τον διαθρωμένο διάλογο στο οποίο ήδη καλέσαμε και την πρόεδρο Κώστα. Στα πλαίσια της διάσκεψης για την νεολαία στη Ρώμη, η Ιταλική Προεδρία θέλει να οργανώσει και άλλες συνόδους ε, μελέτης των θεμάτων που βρίσκεται στο κέντρο των τριών προεδριών, το Youth Empowerment, με ειδική έμφαση στην συμμετοχή, την πολιτική συμμετοχή, θέμα που έχει ξεχαστεί κάπως και θέλουμε να ξαναβάλουμε στο κέντρο των συζητήσεων. Τις ίδιες μέρες θα γίνει η συνάντηση των Γενικών Διευθυντών των χωρών της Ένωσης με δύο βασικά θέματα. Πρώτον, την υγεία των, ε, ναι, Υγεία και νέοι με έμφαση στις παθολογικές εξαρτήσεις και την, και την ε, πρόληψή τους και δεύτερον την ε, πολιτική υπηρεσία ιδίως την ιδέα μιας ευρωπαϊκής εθελοντικής πολιτικής υπηρεσίας προς την κατεύθυνση που ανέφερε ο Πρωθυπουργός κ. Ρέντσι όταν μίλησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της παρουσίας της Ιταλικής Προεδρίας τον Ιούλιο. Η εθελοντική αυτή υπηρεσία θα έχει ρόλο και εμπειρία και ηθαγένεια και αστική δέσμευση και προσανατολισμό στις εθελοντικές δραστηριότητε, αλλά ταυτόχρονα και την ευκαιρία αναζήτησης και εντοπισμού του επαγγελματικού δρόμου του καθενός. Δεν είναι τυχαίο ε, ότι η Ιταλία θέλησε να εντάξει την πολιτική υπηρεσία μεταξύ των διαφόρων εναλλακτικών δυνατοτήτων που επιτρέπονται μέσα στο πρόγραμμα εγγύησης νέων, πρόγραμμα που στην Ιταλία ε, είχε μεγάλη επιτυχία. Πάνω από 170.000 άτομα γράφτηκαν ήδη στο πρόγραμμα αυτό. Η Ιταλία έχει διευρύνει το πρόγραμμα αυτό μέχρι την ηλικία των 29, ε, προεξοφρώντας ακριβώς αυτά που, είχαν, ε, που είχε αναφέρει το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 17ης Ιουλίου. Στο χρονοδιάγραμμα της Ιταλικής Προεδρίας ε, υπάρχουν και άλλα ραντεβού. Πρώτον, αυτό της Εθνικής Υπηρεσίας Νέων με τίτλο «Gioventù Ιταλά, Ιταλιάνα, ε, εγγύηση για την Ευρώπη. Θα γίνει στις 5-6 Νοεμβρίου στην ε, Ρώμη και θα εξετάσει και το μέλλον του προγράμματος Erasmus Plus και το μέλλον των, της νέων. Στο Μιλάνο τέλη Οκτωβρίου επίσης γίνεται μια διάσκεψη για το θέμα ε, αναγέννηση της συμμετοχής ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Υπηρεσίας. Εκεί θέλουμε να αναδείξουμε την ε, πρόταση αυτής της Ευρωπαϊκής ε, Εναλλακτικής Πολιτικής Υπηρεσίας Υπάρχει ένα πειραματικό σχέδιο της Κομισιόν Ιταλία, Γαλλίας, μεταξύ Ιταλίας, Γαλλίας και Γερμανίας για την πειραματική χρήση της υπηρεσίας αυτής που δεν έχει αυτή τη στιγμή νομοθετικό πλαίσιο, είναι μια εθελούσια δράση. Ε, μια τελευταία πρωτοβουλία, πάντα από την Εθνική Υπηρεσία Νέων, είναι το Youth Work, μια σύνοδο στις 10 Δεκεμβρίου που θα αναδείξει τις θεματικές της άτυπης και τυπικής ε, εκπαίδευσης για την αναγνώριση των ε, ε, δεξιοτήτων που αποκτώνται έτσι. Κλείνω λέγοντας ότι οι νέοι είναι αυτοί που γεννούν την καινοτομία, αλλά ταυτόχρονα είναι πολίτες του σήμερα, όχι του αύριο. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε πολιτικές νέων που να είναι πραγματικά αποτελεσματικές. Ευχαριστώ τον κύριο Υφυπουργό για την παρέμβασή του που ήταν πλήρης και καλύπτει το θέμα της δημιουργίας μιας πραγματικά ευρωπαϊκής πολιτικής υπηρεσίας. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, όπως ε, και το ότι η διακυβέρνηση των πολιτικών για τους νέους να γίνεται σε ευρωπαϊκό και όχι σε εθνικό επίπεδο. Οι συνάδελφοι που θέλουν να λάβουν το λόγο. Παρακαλώ. Καταρχάς ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, μια σύντομη παρατήρηση καταρχάς. θυμάμαι ε, ιδιαίτερα ε, κατά τη διάρκεια της ε, Πολωνικής Προεδρίας τι δύσκολα χαρακτήρα έχει όλη αυτή η εργασία. Η Προεδρία όμως των έξι μηνών είναι πάρα πολύ σύντομη και έτσι δυστυχώς δεν υπάρχει ο επαρκής χρόνος για να κληρωθούν όλες αυτές οι πρωτοβουλίες που παρουσιάζει κάθε Προεδρία. Ιδίω ε, στο θέμα του αθλητισμού των νέων πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προτεραιότητα ε, και να συμπεριλάβουμε όλους τους νέους. Ε, οι ιδέες σας είναι πάρα πολύ θετικές και πιστεύω ότι πρέπει και εμείς να συνεχίσουμε, να υποστηρίξουμε τις ε, πρωτοβουλίες που ήδη λειτουργούν, που ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή, έχουν ξεκινήσει και ε, δεν είναι καθόλου αρνητικό να η ντροπή να συνεχίζουμε ε, παρελθούσες δράσεις και, να συνεχίσουμε σε, προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα λοιπόν να εκμεταλλευτούμε και να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα οποία ήδη γίνονται, εξελίσσονται. Δεύτερον, ε, να δώσουμε ε, την ευκαιρία σε όλα τα κράτη να ενισχύσουν αυτούς τους τομείς ε, των νέων του αθλητισμού. Και ελπίζω ότι και εσείς κύριε Υπουργέ θα μπορέσετε να εξασφαλίσετε αυτά τα προγράμματα και χρηματοδοτικά με τις απαραίτητες πιστώσεις και τρίτον ο αθλητισμός είναι βέβαια ένα πάρα πολύ καλό στοιχείο και για την φυσική ευρωστία, όμως πολλές φορές οδηγεί και σε ε, τραυματισμούς ή ατυχήματα, ιδίως στους νέους. Θα ήθελα λοιπόν στην Ευρώπη να γίνει μία συζήτηση για τους νέους αθλητές που αναγκάζονται ε, πολλές φορές και κάτω των, όταν είναι νεότεροι από 18 ετών ε, να παραιτηθούν από τον αθλητισμό λόγω τραυματισμού ή άλλων ατυχών γεγονότων. Οι νέοι αυτοί ε, θυσιάζουν πάρα πολλά, αφιερώνονται στον αθλητισμό και πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε όταν πλέον σταματήσει η εξέλιξή τους, η καριέρα τους. Είναι ένα μικρό παράδειγμα αυτό. Ε, θα ήθελα να ε, συνεχίσουμε λοιπόν τις καλές πρωτοβουλίες που ήδη έχουν ξεκινήσει στην Ευρώπη και να μην ε, αποκλείσουμε τις ενέργειές μας σε μεμονωμένα γεγονότα ή τομείς. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, Παίρνω το λόγο, διότι όπως και ο συνάδελφος που μόλις μίλησε, πιστεύω ότι δεν υπάρχει πολύ χρόνος για μια προεδρία για να δράσει. Αλλά γι' αυτό το λόγο είναι ακόμη πιο σημαντικό όταν μια χώρα έχει την Προεδρία και αποφασίσει να επεξεργαστεί επίμονα ένα θέμα, να το προωθήσει. Αυτό το θέμα θα μπορούσε να είναι ενδιαφέρον και για το μέλλον, όχι μόνο για μία Προεδρία είναι σημαντικό να χτίζουμε κάτι και για το μέλλον. Τι θέλω να πω με όλα αυτά. Κύριε Μπόμπα, αντιλαμβάνομαι πόσο αποφασισμένος είσαστε και είμαι σίγουρος ότι αυτό δεν αφορά μόνο την περίοδο της προεδρίας σας. Οπωσδήποτε θα ακολουθήσετε την ίδια γραμμή και μελλοντικά. Αλλά θέλω να συζητήσω το θέμα των ικανοτήτων και την προώθηση των δικαιωμάτων των νέων και την πρόσβαση σε αυτά τα δικαιώματα. Όπως είπατε πολύ σωστά, είναι πολίτες του σήμερα και όχι του μέλλοντος οι νέοι. Στην Ευρώπη έχουμε ασχοληθεί πολύ με το θέμα της απασχόλησης των νέων. Πιστεύουμε λοιπόν ότι πολλά πράγματα θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί τον κύριο Μπόμπα βέβαια, αλλά και με τον κύριο Γιούγκερ πρέπει να συζητήσουμε. Δηλαδή να τον ρωτήσουμε πώς θα εφαρμόσει αυτά που πρέπει να εφαρμοστούν για τους νέους και τα έχουν υποσχεθεί όλοι προεκλογικά. Έχουμε λοιπόν τη δημόσια υπηρεσία, την ευρωπαϊκή. Ωραία θέλουμε να δούμε να εξελιχθεί αυτή η υπηρεσία. Ουσιαστικά. Σας ευχαριστούμε για όσα είπατε και ελπίζουμε να επιμείνετε προς την ίδια κατεύθυνση. Ευχαριστώ που ε, παρουσιάσατε κι εσείς τις προτεραιότητες της Ιταλικής Προεδρίας των τομέα των νέων, έχω μία παρατήρηση και, ένα, και μία ερώτηση. Είναι σημαντικό να υποστηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση την ενεργό συμμετοχή των νέων ως πολιτών για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την, ε, το σεβασμό όλων των δικαιωμάτων τους και να μπορούν και εκείνοι να ενεργούν υπεύθυνα. Ορισμένες φορές οι νέοι δεν χρησιμοποιούν το δικαίωμα της ψήφου ε, όσο θα μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν και έτσι θα πρέπει να ανταποκριθούμε στις ανάγκες τους. Αλλά ε, πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Οι πολιτικοί σε όλες τις χώρες πρέπει να έχουν κατά νου ε, τις ε, ανάγκες των νέων, ιδιαίτερα στην οικογενειακή πολιτική και βέβαια στην πολιτική της απασχόλησης. Γι' αυτό υποστηρίζω θερμά την παροχή πιστώσεων, των αναγκαίων πιστώσεων στην παιδεία και ιδίω ε, σε αυτήν που απευθύνεται στους νέους, διότι έχει τεράστια ωφέλη. Και μία ερώτηση τώρα, κύριε Υπουργέ, όσον αφορά τις εγγυήσεις στους νέους. Υπάρχει ένας περιορισμός παροχής πιστώσεων στις πιο επικίνδυνες, στους πιο επικίνδυνους τομείς όπου η ανεργία είναι πάνω από 23%. Σε ορισμένε περιπτώσεις μπορούμε να ανεβάσουμε το επίπεδο πέραν των 25 ετών, αναφέρεται εσείς 29. Ότι το έχετε εφαρμόσει στην Ιταλία και ότι μπορούν να υποφεληθούν από τις υπάρχουσες πιστώσεις ε, ε, και μετά τα 25. Είπατε όμως ότι μπορεί ενδεχομένως να παρασχεθεί η εγγύηση αυτή ακόμα και σε τομείς όπου η ενεργεία δεν είναι άνω του 23%. Αυτό μπορεί ίσως να γίνει σε ορισμένες χώρες, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες η Πρόεδρος. Η κυρία Τινόλφη, με την ευκαιρία της παρουσίας ε, του Υπουργού, θέλω να θέσω μια ερώτηση στον κύριο Υφυπουργό. Τι έγινε πέραν του site και της καταχώρησης για την εγγύηση των νέων. Στην προηγούμενη συνάντηση μας είπατε ότι στην Ιταλία το πρόγραμμα ξεκίνησε 1η Μαΐου. Τέσσερις μήνες και δύο μέρες δηλαδή. Έκτοτε. Σε αυτό το τετράμινο πόσοι νέοι βρήκαν δουλειά όπως προβλέπει το πρόγραμμα. Για να δώσουμε συγκεκριμένα στοιχεία στην Ευρώπη. Και μετά συνεχίζει, πτηρεί το πρόγραμμα αυτό τις προσδοκίες που έχουν δοθεί να βρουν δηλαδή οι δραστηριότητες ή τι γίνεται για να μειωθούν τα προβλήματα αν τυχόν υπάρχουν προβλήματα. Η κυρία Ward. Ευχαριστώ. Όλη μου τη ζωή εργάστηκα μαζί με νέους στον τομέα της τέχνης, του πολιτισμού και προσπάθησα να, να προσφέρω ε, την κατάλληλη κατάρτιση, δεξιότητες. Πιστεύω ότι πρέπει οι νέοι να έχουν ε, λόγο στη λήψη των αποφάσεων και το μέλλον πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώνουν και εκείνοι το μέλλον τους. Αναφερθήκαμε στις καινοτομίες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για να έχουμε καινοτομίες θα πρέπει οι πολίτες να έχουν ένα ασφαλές περιβάλλον μέσα στο οποίο να μπορούν να αναλαμβάνουν κινδύνες, το ρίσκο να προσφέρουν κάτι καινούριο και ιδίως ως καλλιτέχνες έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις πρωτοβουλίες τους. Δεν ασχολούμαι τόσο πολύ με τον αθλητισμό, αλλά πιστεύω ότι με την τέχνη μπορεί κανείς να ενδυναμώσει, να ενθαρρύνει τους νέους ε, και να τους βοηθήσει να συμμετέχουν, να συμμετάσχουν και αυτοί στη διαμόρφωση του μέλλοντός τους. Νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Μπόμπα για να απαντήσει. Ένα ερώτημα για τον αθλητισμό ήταν. Πιέζω γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις και τα ερωτήματα. Προς τον συνάδελφο Στροβιεύσκη. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Η Προεδρία κρατάει λίγο, έξι μήνες. Δεν χρειάζεται να δημιουργήσουμε τίποτα εκ του μηδενός. Άρα είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε ε, νόημα στην ε, συνέχεια των πολιτικών. Δίνουν αποτελέσματα δηλαδή. Δεν μπορούμε να μειώσουμε τις πολιτικές ε, μόνο στα γεγονότα. Η Ιταλική Προεδρία λοιπόν σε ό,τι αφορά την πολιτική νέων θέλει να επικεντρώσει την προσοχή της σε δύο θέματα. Ένα που ισχύει στις ευρωπαϊκές πολιτικές, την εγγύηση νέων, να γίνει μια διαθροτική, συνεχιζόμενη, συνεχής πολιτική και όχι μόνο για ένα-δύο χρόνια όπως προβλέπετε τώρα, να γίνει ένα διαθροτικό στοιχείο, ώστε όλοι οι νέοι που δεν έχουν δουλειά, ούτε εκπαίδευση να έχουν μια ευκαιρία να προσεγγίσουν, να μάθουν, να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Και το δεύτερο, το θέμα που ανέφερα προηγουμένως, της ε, πολιτικής υπηρεσίας, ούτε και εδώ δημιουργούμε κάτι από τις καλύτερες εμπειρίες που έχουμε στις διάφορες χώρες ε, και μίλησα για το πιλωτικό σχέδιο της Επιτροπής να δούμε αν η προοπτική αυτή της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Υπηρεσίας μπορεί να γίνει ένα από τα στοιχεία που θα ε, επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε την κουλτούρα και τους δεσμούς των νέων στην Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά την συνάδελφο Μόργαν, συμφωνώ μαζί της. Πιστεύω ότι το θέμα της πρόσβασης στα δικαιώματα είναι ουσιαστικό, δηλαδή παρέχει ευθύνες. Δεν είναι... Δεν πρέπει να βλέπουμε τους νέους ε, σαν να είναι μακριά από την πραγματικότητα. Η ευθύνη αυτή θα πρέπει να παρέχεται και μέσω αυτού να αποκτά ε, πρόσωπο και η καινοτομία και κοινωνικά και πολιτικά για τη συνάδελφο Σοϊντρόβα. Συμφωνώ ότι οι πολιτικοί πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι νέοι σε πολλές χώρες έχουν ε, ποσοστό συμμετοχής, ε, ε, συμμετοχής σε εκλογές χαμηλότερο από άλλα τμήματα του πληθυσμού. Αυτό είναι ένα καμπανάκι που πρέπει να μας ξυπνήσει. Όποιος κάνει πολιτικές δραστηριότητες και γνωρίζει την περιοχή ε, το χώρο στον οποίο δουλεύουμε, πρέπει να το παρακολουθήσουμε προσεκτικά. Είναι ένα μήνυμα ότι ε, φτωχαίνει η δημοκρατική διαδικασία αν οι νέοι δεν ε, καταλαβαίνουν τη σημασία της δημοκρατίας. Αυτό δεν θα μπορέσει να επιτρέψει, δεν θα επιτρέψει να αλλάξει και την ε, και τη δική μας ε, ευθύνη σε αυτό. Σε ό,τι αφορά το θέμα εγγύησης νέων, δεν νομίζω ότι υπάρχει το όριο του 23% πρόσβαση στο πρόγραμμα. Μετέχουν στο πρόγραμμα όλοι οι νέοι που δεν ε, είναι σε θέση εργασίας ή δεν είναι σε κάποια μορφή εκπαίδευσης. που βρίσκονται σε μια κατάσταση αβέβαιη μεταξύ δουλειά και εκπαίδευση. Η Ιταλία πέρασε την ηλικία στα 29 και είδαμε με χαρά ότι το Κοινοβούλιο υιοθέτησε ένα ψήφισμα που πηγαίνει προς την ίδια κατεύθυνση. Νομίζω ότι ο προσανατολισμός αυτός θα πρέπει να είναι ένας προσανατολισμός που θα πρέπει να υιοθετηθεί γενικότερα. Σε ό,τι αφορά την κυρία Ντινόλφη νομίζω ότι είναι πρόημο, δεν ξέρω τα στοιχεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και στην Ιταλία νομίζω ότι είναι πρόημο να ε, προσπαθούμε να, κρίνουμε ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε πριν από λίγους μήνες και που ε, περιλαμβάνει σημαντική εμπλοκή και της ε, κυβέρνησης. Τέλος του 2015 θα έχουμε τις, τα πρώτα αποτελέσματα όταν, όταν αποδεσμευτούν όλοι οι πόροι. Τέλος, ό,τι αφορά το ερώτημα της κυρίας Word, νομίζω ότι η επιλογή πρέπει να είναι της διεύρυνσης των ευκαιριών και δυνατοτήτων, αλλά και του χώρου ε, ψυχαγωγίας και κοινωνικονομικής και κοινωνικοεκπαιδευτικής κατάρτισης των νέων θα είναι να επιτρέψουμε να, να χρησιμοποιηθούν αυτές τις δυνατότητες για την ανάπτυξη των νέων και επαγγελματικά και οικονομικά. Προς την κατεύθυνση αυτή ο διαθωμένος διάλογος θα πρέπει να μας οδηγήσει στον εντοπισμό καλύτερα των ε, δυνατοτήτων που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη αυτή σε ένα προστατευμένο κατά το τρόπο περιβάλλον που θα επιτρέψει ωστόσο στους νέους να έχουν μια γενικότερη ευθύνη ενώπιον έναντι της κοινωνίας. Για τον αθλητισμό θέλετε να πείτε κάτι. Δύο λεπτά όμως. Γιατί έχουμε λίγο χρόνο και συντονιστές μετά. συνοπτικά το πρόγραμμα της Προεδρίας για τον αθλητισμό. Πρώτον, να ενεργοποιήσουμε ό,τι εγκρίθηκε χάρη στη δουλειά της Ελληνικής Προεδρίας στο πρόγραμμα εργασίας που αφορά το 2014 2014-2017. Ε, Δεύτερον, η Προεδρία θεωρεί πολύ σημαντικό το θέμα της του αθλητικού, της αθλητικής κουλτούρας ως στοιχείο κοινωνικής ένταξης και θα δώσει μεγάλη σημασία σε αποτελεσματικές σχέσεις για την καταπολέμηση της, των στημένων αποτελεσμάτων, των στοιχημάτων. Νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Ε, το πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικές εκδηλώσεις, ιδίως μια συνάντηση των Υπουργών Αθλητισμού στη Ρώμη 20-21 Οκτωβρίου, Συμβούλιο Υπουργών 25 Νοεμβρίου και διαρθρωμένος διάλογος για τον αθλητισμό με γεύμα εργασίας στις 25 Νοεμβρίου. Η Προεδρία κατόπιν θα ασχοληθεί με άλλα δύο σημαντικά ειδικά θέματα, την έκθεση, τη σχέση μεταξύ αθλητισμού και καινοτομίας. Σε πολλές περιπτώσεις οι νέες τεχνολογίες μπορούν να δώσουν σημαντική, έχουν σημαντικές επιπτώσεις. Και κάτι πολύ σημαντικό είναι προσοχή στην ανάπτυξη της ε, αθλητικής ε, άσκησης για να υπογραμμίσουμε την, ε, τα, θεων, τα, τα πλεονεκτήματα για την υγεία, ιδίως σε σχολική και νανική περίοδο. Και κάτι πολύ σημαντικό, τα τελευταία στοιχεία μας λένε ότι η πρακτική αυτή, η άσκηση μειώνεται, ενώ αυξάνονται οι καθιστικές μορφές ζωής και η ε, παιδική παχυσαρκία, ανησυχητικά μάλιστα. Η χρήση λοιπόν των σχολείων και των ενώσεων αλλά και της ε, εξωσχολικής δραστηριότητα είναι πολύ σημαντική για το ερώτημα που θέσατε θα δώσω το λόγο στον κύριο Πανεμπιάνκο. Ευχαριστώ. Εντάχει κι εγώ. Να συμπληρώσω αυτά που είπε ο Υφυπουργό για τον κεντρικό χαρακτήρα του αθλητισμού και τις σχέσεις αθλητισμού σχολείου. να τονίσω ότι υπάρχει προσοχή της Ιταλικής Προεδρίας στο θέμα αυτό. Επίσης, στον τομέα αυτό δώσαμε προσοχή σε σχέση ιδίως με μια ειδική ε, ρύθμιση για τα αθλητικά λύκεια. Ένα ειδικό χώρο στον οποίο θα ενσωματώσουμε την σχέση σχολειο αθλητισμού. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα ε, για την Ιταλική Προεδρία. 20 και, 13, 20, ε, και 12 και μέχρι 13 ε, Σεπτεμβρίου θα γίνει στην Ιταλία μια, ε, μια συνέλευση για αυτό το, το ζήτημα ακριβώς. δηλαδή το, το διπλό, το σχολείο και τον αθλητισμό και μια εκδήλωση για το ΕΑΣ, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο. Νομίζω ότι Καιρό να σταματήσουμε εδώ. Θα ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Πρεδρία για την παρουσία τη. και να υπενθυμίσω ότι και η πρόσφατη έκθεση που εγκρίναμε, μάλλον όχι πρόσφατη, που εγκρίναμε πριν από δύο χρόνια, περίπου, χρόνια περίπου για τον αθλητισμό και την ανάγκη να γίνει ε, αρμοδιότητα της Ένωσης, κάλυπτε και το θέμα της διπλής σταδιοδρομίας, δηλαδή του αθλητικού σχολείου. Να ήρθε ο κύριος Φίσας. Ε, αυτό έλεγα τώρα για σας για την έκθεσή σας κύριε Φίσας. Σταματώ εγώ εδώ. Το Κοινοβούλιο ζήτησε να επεκταθεί στα 29 η εγγύηση νέων. Ελπίζω να είναι επόμενη απόφαση. Η Ιταλία σας θυμίζω ότι μετά το 2015 θα πρέπει να ξαναχρηματοδοτηθεί η εγγύηση νέων δεν θα έχετε την προεδρία τότε, αλλά πραγματικά είναι σημαντικό να αναχρηματοδοτηθεί η εγγύηση νέων για το μέλλον. Σας ευχαριστώ. Πιστεύω ότι μπορούμε να χαιρετήσουμε τους ε, προσκεκλημένους μας. Και ζητώ να φύγετε όλοι. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Έχουμε εντάχει μια διάσκεψη, ε, μια συνάντηση συντονιστών για 20 λεπτά περίπου. Φύγετε γρήγορα αν γίνεται.